Buongiorno a tutti. Καλημέρα σε όλους σας. Yes. Now we start. Yeah. Punto 11, no? Niente là, Sandra. Buongiorno a tutti, Καλημέρα σε όλους σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα αρχίσουμε άμεσα με την ψηφοφορία. Γι' αυτό ζητώ από όλους τους συναδέλφους να μου πούνε αν έχουν μαζί τους την κάρτα ψηφοφορίας τους. Σημείο 11 της ημερησίας διατάξεως, θέσπιση του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Παρέρε Σάντρα Κανιέτε. Σάντρα Κανιέτε, η συντάκτρια γνωμοδότηση. Σάντρα, θέλεις να πάρεις το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα για να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συμμετείχουν στην ε, ε, εκπόνηση της γνωμοδοτήσεως αυτής έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ορθό και ισορροπημένο. Είχαμε πάρα από 100 τροπολογίε και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Molto bene, grazie Sandra. Ευχαριστώ πολύ Σάντρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχετε βάλει ήδη το, την κάρτα της ψηφοφορίας σας. Άρχεται η ψηφοφορία επί του άρθρου 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν έχετε την κάρτα σας. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το σημειώνουμε. Εψήφισαν όλοι υπέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Mm? Eh, ο αντιπρόεδρο Παπαστάνκο, εάν συμφωνείτε όλοι, ζητάει αν μπορούμε να ψηφίσουμε on μπλοκ. Γιατί σε όλα έχουμε θετική γνωμοδότηση τη εισηγητρία, σε όλε τι τροπολογίε αυτέ. Είναι δυνατόν, πιστεύετε, όχι, θέλετε, υπάρχει κάποια διαφορετική ψηφοφορία. Πέστε μας στη δικιά μας περίπτωση έχουμε και κάποιες αρνητικές ψηφοφορίες. Μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι την 26, αν θέλετε, on block. Όχι, ούτε αυτό δεν γίνεται. Ακούγονται φωνές διάφορες. Εντάξει, μία-μία τις τροπολογίες λοιπόν. Να ψηφίσουμε διανατάσσεως της χειρός. Όχι, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Σιλβέστρες. Εάν οι άλλε ομάδε έχουν μία ή δύο αρνητικέ ψηφοφορίε, ενώ το ΕΛΚΑ έχει μόνο θετικέ, να ψηφίσουμε πρώτα αυτέ τι τροπολογίε επί των οποίων υπάρχει αρνητική θέση και μετά να κάνουμε unblock τα υπόλοιπα και να τελειώσουμε πολύ γρήγορα. Ωραία. Διανατάσσεω τη χειρό λοιπόν. Το 15 το ψηφίσαμε ήδη. 16 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Τρει. 3 τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 Νεντελτσέβα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 21 καρόνα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 Σιλβέστρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 Γκέρλινγκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε 24-25 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά αποχέσε εγκρίνεται. 29 υπέρ. 29 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Όχι, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 29 άρχεται η ψηφοφορία.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 42 υπέρ, υπέρ τη 42 κατά. Εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 4 υπέρ, κατά. αποχέ. εγκρίνεται. 45 Ρέιμερς. Όλοι υπέρ του 45. Κατά. Μήπως εδώ να κάνουμε επαλήθευση. Ωραία, επαλήθευση από τις τροπολογίες 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. «46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 θαύρο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 Ρέιμερς υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 και εδώ εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται με την ίδια, τροπολογία, ε, με την ίδια πλειοψηφία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 58 σιλβέστρες υπέρ κατά εγκρίνεται. Ε, έλεγχος, ωραία, όχι. Έχουμε τώρα τις αιτιολογικές σκέψεις. Να ψηφίσουμε αν μπλοκ τις αιτιολογικές σκέψεις, όχι. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 6 Σικερέσκι. πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται, εγκρίνεται ε, υπερθυμών 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένα εισηγητής του εισηγητού μάλλον υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 8 Σικερέσκη. υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 9 υπέρ κατά κατά με ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται Υπαριθμόν 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2 της ήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 11. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 12. Το 11 θέλετε. 11, 11, 11, εντάξει. Να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 11. Εψήφισαν όλοι ηλεκτρονική επαλήθευση για το 11. Απορρίπτεται. Είχατε δίκιο. 12 τώρα. Μπρίτα, θες να πεις κάτι? Όχι. 12 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14 Τέλος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται κατά την άποψή μου, λέει ο Πρόεδρος. Τελική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση έτσι όπως έχει ε, τροποποιηθεί, αλλά θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία λοιπόν, επί του τροποποιημένου κειμένου, ψήφισαν όλοι. Άψογα και εγκρίνεται ε, συγχαρητήρια Σάντρα Καλνιέτε. Σημείο 12. Ειδικό πρόγραμμα υλοποίηση προγράμματος ε, ε, έρευνα και καινοτομία ορίζον 2020. Ξανά είναι η συγγήτρια η Σάντα Καλνιέτε. Εάν δεν θέλετε να πάρετε το λόγο μπορούμε να ξεκινήσουμε απευθείας. Συνεχίζουμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία 8, Σικιέρσκι. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εδώ μου φαίνεται ότι παίζεται στην ψηφό, εγκρίνεται. Πάντοτε Υπέρ της 9. Υπέρ κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 9. Άρχισε η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Υπέρ της 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές δεν περνάει. Αποχές εγκρίνεται. 18-19 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. απορρίπτεται υπέρ της 20 κατά αποχές εγκρίνεται όχι ελέγχουμε 20 Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι για την 20. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την Κίρλινγκ. Ψηφίσατε όλοι για την 21 απορρίπτεται. 23 υπέρ υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Ναι, δίκιο έχετε, απορρίφθηκε. Υπέρ της 24, Γέρλινγκ, υπέρ κατά αποχές, κατά, κατά, εγκρίνεται. 25, υπέρ της 25, κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται 41 σκοτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 3 Σικέρσκι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε θα έλεγα απορρίφθηκε απορρίφθηκε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία της ε, νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ωραία. Συγχαρητήρια στη Σάντρα Κανιέτε. Σημείο 13. Σημαντικό νέο. Συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα. Η Ράτσε Γκαρσία Περές τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου. Τα επόμενα δύο σημεία αφορούν στα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα και στους κανόνες εμπορίας και αποτελούν μέρος του ιδίου πακέτου με την ίδια εισηγήτρια, την κυρία Γκαρσία Περές. Ένας τρίλογος έγινε στις 21 Ιουνίου και μετά από την επιτυχία της διαπραγμάτευσης καταφέραμε έναν συμβιβασμό με το Συμβούλιο. Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας της 25 Ιουνίου ενέκρινε μία νέα μόνιμη πλέον έκδοση του κανονισμού που μοιράστηκε και θέλουμε να πάμε στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο με το θέμα. Λοιπόν, μπορεί τώρα να μας πληροφορήσει για όλα τα πακέτα η Ράτσε. Πάρα πολύ σύντομα για να πω Μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων και τριλόγου σχετικά με αυτό το κανονισμό για τα συστήματα ποιότητας, Κάναμε το τεστ για το νέο ρόλο του Κοινοβουλίου, όπως προκύπτει μετά από τη Λισαβόνα. Και φάνηκε ότι και το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να το έχουν καθαρό, ότι το Κοινοβούλιο σήμερα μετράει και ότι πρέπει να λάβουν οπωσδήποτε υπόψη τους ε, τη δουλειά αυτής της Επιτροπής. Εμείς ε, είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς. Τώρα ένα από τα ουσιαστικά ζητήματα τα οποία υπήρχαν στο τραπέζι από το Κοινοβούλιο, δηλαδή το θέμα του όγκου παραγωγής από τις οργανώσεις παραγωγών, αυτό δεν πέρασε μέσα στα άρθρα του κανονισμού. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει μία δήλωση εκ μέρους του Συμβουλίου όπου γίνεται αναφορά σε αυτό το θέμα σχετικά με τις ομάδες παραγωγών ότι το Κοινοβούλιο ναι καταλαβαίνει τη θέση του Κοινοβουλίου και καταλαβαίνει ότι στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα πρέπει να ληφθεί αυτό το στοιχείο υπόψη. Επέμεινε λοιπόν για αυτή την πολιτική δήλωση. Εμείς δεν ε, ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά τουλάχιστον γίνεται σχετική αναφορά. Για τα υπόλοιπα θέματα καταφέραμε να καταλήξουμε σε το οποίο γίνεται καθαρό όλο το θέμα των διαδικασιών, το θέμα της απλούστευσης των συστημάτων ποιότητας, ενίσχυση του ρόλου των ομάδων παραγωγών, ζητήματα που για μας ήταν σημαντικά, όπως ο καθορισμός πλέον του ε, προϊόντος ε, ε, ορεινής προέλευσης για την απευθείας πώληση και εκεί έχουμε μία αναφορά και ζητούμε από την Κομισιόν να μας παρουσιάσει μία μελέτη σχετικά συμπεριλαμβάνοντας και όρους ε, ποιότητας ε, για νησιωτικά προϊόντα ή άλλα σχετικά με, τις ε, παραδοσιακές, με τα παραδοσιακά εγγυμένα προϊόντα οι Βρετανοί και οι Ανατολικοί συνάδελφοι πρέπει να είναι ευτυχείς διότι καταφέραμε να πετύχουμε να περάσουμε τη θέση μας, δηλαδή τον συμβιβασμό που πετύχαμε σε αυτήν την Επιτροπή, να μείνει δηλαδή το status quo. Τώρα για άλλα ζητήματα διαδικαστικά πέρασαν αυτά που ήθελε το Κοινοβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω για την τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία των σχεδόν εισηγητών από όλες τις πολιτικές ομάδες. Εγώ θέλησα να λάβω αποφάσεις συλλογικά και να λάβω υπόψη τις θέσεις όλων των συναδέλφων. Τους ευχαριστώ για την παρακολούθηση αυτού του ντοσιέ. Θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία της ε, Επιτροπής, αλλά και του συνεργάτες μου, του γραφείου μου, που με βοήθησαν. Ήταν μια μακρόπνοη εργασία, καταφέραμε όμως να έχουμε το αποτέλεσμα που η παραγωγή προϊόντων ποιότητες ε, ε, θέλανε. Και ελπίζουμε τον Σεπτέμβριο να έχουμε την επισφράγηση όλης αυτής της εργασίας. Ε, ευχαριστώ Ιράτσε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν πετύχαμε το 100% αλλά τουλάχιστον πετύχαμε το 90%. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτά τα οποία δεν πετύχαμε, δηλαδή την επέκταση του, του προγραμματισμού παραγωγής και με τη θέση που ο Βισελ Νταντέν έχει αναλάβει μέσα στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ, ε, θα, θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε. Είναι σημαντικές οι αλλαγές που επέφερε το Κοινοβούλιο σε αυτό το κείμενο. Άμα συγκρίνεται την πρόταση της Κομισιόν και το τελικό κείμενο που έχετε μπροστά σας θα δείτε ότι μοιάζουν ελάχιστα μεταξύ τους. Και αυτό οφείλεται στην δουλειά του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής μας και της εισηγήτριας. Ο Σμιθ ζήτησε το λόγο. Η, συγγνώμη Σμιθ, η Ράτσε. Να τονίσω κάτι που ξέχασα. Ήθελα να πληροφορήσω στην Επιτροπή μας ότι τον Σεπτέμβριο θα ψηφίσουμε μόνο τα συστήματα ποιότητας. Οι προδιαγραφές του μάρκετινγκ θα ξέρετε ότι δεν έχει καν ξεκινήσει διαπραγματευτική εντολή από το Συμβούλιο. Οπότε αυτό δεν θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Ναι, ναι, πολύ καλή διευκρίνηση. Ο Σμίθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι αν έπρεπε να είμαι θυμωμένο σήμερα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί θυμωμένοι Βρετανοί, οπότε δεν υπάρχει λόγος να θυμώσω κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, να συγχαρώ την Ιράτσε, ε, γιατί δούλεψε πάρα πολύ καλά σε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα και συνεργάστηκε πολύ καλά με τους ε, συναδέλφους ε, και νομίζω ότι και εκείνη και η ομάδα της και η γραμματεία ε, χαίρουν, αξίζουν συγχαρητήρια γιατί πραγματικά δούλεψαν πάρα πολύ καλά σε ένα δύσκολο θέμα. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ρεαλιστές σχετικά με αυτά που επιτύχαμε και εν πάση περιπτώσει καταφέραμε ε, να πείσουμε το Συμβούλιο να κάνει πράγματα τα οποία δεν ε, ήθελε. Καταφέραμε κάποια πράγματα όσον αφορά τους πολίτες ε, και τους παραγωγούς, αλλά δυστυχώς δεν πλησιάσαμε καν τους τα στοιχεία τα οποία είχαμε θέσει εμείς σαν προϋποθέσεις και σαν στόχους ε, για την ε, Επιτροπή μας εδώ. Εν πάση περιπτώσει, χρήσιμα αυτά που αναφέρονται για τις εγγυημένες τοπικές παραγωγές ε, και για τα ορεινά προϊόντα. Τώρα, η αξία μιας πολιτικής δήλωσης είναι γνωστή, την ξέρουμε, αλλά νομίζω ότι εδώ δεν είχαμε και πάρα πολύ βάρος στην προκειμένη περίπτωση. Ε, Βεβαίω η πολιτική είναι η τέχνη του ε, εφικτού, ε, και, αλλά καμιά φορά τα μαθηματικά είναι ε, εναντίον μας. Να μην γελιόμαστε πάντως, να μην γελιόμαστε. Βλέποντας το άρθρο για την Agro Europe, εκεί όπου είπατε κι εσείς ότι η ε, συμφωνία αφορά απόδειξη της ε, προστιθέμενης αξίας. Τι να σας πω, εγώ δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος ότι έτσι είναι. Ε, ξέρουμε ότι και στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις ε, τα διακυβεύματα είναι μεγάλα. Δεν ξέρω κατά πόσον θα πλησιάσουμε στους στόχους μας. Ε, ε, φαντάζομαι ότι σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσουμε πάλι μέσω συμβαστικών λύσεων. Πάντως η ομάδα μου δεν συμφωνεί με όλους τους συμβασμούς. Ευχαριστώ, συνάδελφε Σμίθ, λέει ο Πρόεδρος. Συμφωνώ καταρχάς με αυτό που λέει ο συνάδελφος Σμίθ, αλλά υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος είναι πολύ σημαντικός τα και θα το πει και ο Ντόρφμαν σε λίγο. Για τα ορεινά προϊόντα υπάρχει η ε, ρητή ε, υποχρέωση αφαίρεσης των προϊόντων, τα απομάκρυνση των προϊόντων, τα οποία καταχρηστικά χρησιμοποιούν ε, την εγγυημένη ονομασία. Ο συνάδελφο Ντόρφμαν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Ιράτσα για τη δουλειά που έκανε. Νομίζω ότι αυτούς τους τελευταίους μήνες συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά έτσι ώστε να βρούμε μια κοινή θέση για το Κοινοβούλιο που τελικά ε, βοήθησε σε πολλά θέματα επί των οποίων είχαμε επιτυχία. Από αυτή την άποψη δεν καταλαβαίνω τώρα την θέση των πρασίνων, γιατί κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ε, δεν ε, διεφαίνεται η θέση τους να είναι αυτή που τελικά φαίνεται να είναι τώρα. Θα δούμε τώρα στην ψηφοφορία. για να ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση. Το θέμα της ε, προγραμματικής, του ε, ε, παραγωγικού προγραμματισμού, όντως, εκεί κάναμε μόνο ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός και ευελπιστώ ότι στην έκθεση του συναδέλφου Μισελ Νταντά θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. και άλλωστε και το Συμβούλιο πρέπει να καταλάβει ότι ο προγραμματισμός είναι χρήσιμος για τους ε, παραγωγούς. Νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Κατά τα λοιπά, η πολιτική μου ομάδα συμφωνεί με όλα τα όσα επιτύχαμε. Ευχαριστώ πολύ, Χέρμπερτ. Ο Σέρφο Σμίτ ξαναζήτησε το λόγο και μετά η Μπριτάιμερς θα είμαι σύντομα, αλλά δεν μπορούσε να περάσει αυτό ασχολίαστο. Η ομάδα μου δεν άλλαξε καθόλου θέση στη διάρκεια όλων ε, των ε, συναδέλφων. Αν δεν μπαινοβγαίνανε ίσω μερικοί στην αίθουσα θα είχαν καταλάβει ποια ήταν η, θέση τη ομάδα μα. Δεν είναι καινούρια, πάντα η ίδια ήταν. Ευχαριστώ, Μπρίτα Ρέιμερ. Και μετά ε, θα δώσω τον λόγο στο Γενικό Διευθυντή τη Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια η οποία έκανε πολύ σοβαρή δουλειά που δεν ήταν πάντοτε εύκολη διότι φτάσαμε σε σημείο ρήξεως πολλές φορές ήταν πολύ δύσκολη η δουλειά της είχε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και ελπίζουμε ότι θα υπερψηφίσουμε το ε, αποτέλεσμα του τριλόγου και θέλω να κάνω κι άλλη μία παρατήρηση. Εδώ έχουμε μόνο την εξέτηση ενός τμήματος του θέματος, το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί καθ' ολοκληρία κάποια στιγμή. Ευχαριστώ ε, και τώρα ο Γιάννος Πλέμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζει η Κομισιόν την ε, ε, συμφωνία ε, και την έκβαση του τριμερούς διαλόγου έτσι όπως επικυρώθηκε την 25η Ιουνίου. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως την εισηγήτρια για τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων καθώς επίσης και την επικοδομητική προσέγγιση των σκιωδών εισηγητών. Θα ήθελα επίσης να αναγνωρίσω και την σκληρή δουλειά ε, όλων των βοηθών και της, ε, του προσωπικού της ε, γραμματείας. Νομίζω ότι τώρα έχουμε ένα ικανοποιητικό και καλά ισορροπημένο συμβιβασμό. Όσον αφορά τον μελλοντικό κανονισμό για τα προγράμματα ποιότητας, θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας στην, ε, ε, χαίρομαι που η Επιτροπή Γεωργίας ενστερνίστηκε την χρήση των PGOs και PGIs ε, που, και ξέρετε ότι πολλές δραστηριότητες ομάδων παραγωγών έχουν πλέον αναγνωριστεί. Επίσης, ε, το πρόγραμμα αναγνώρισης ε, ποιοτικών προϊόντων και εγγύησης ε, του ονόματος που πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς επιφύλαξη είναι κάτι θετικό. Το Optional Quality Scheme όσον αφορά τα προϊόντα των ορεινών περιοχών ταυτίζεται με τα όσα είχε ζητήσει η Επιτροπή Γεωργίας. Τέλος, όσον αφορά την ευθυγράμμιση του ε, πακέτου ποιότητας ε, με την Λισαβόνα και αυτό έλαβε χώρα. Βεβαίως, η ε, η ποικιλότητα των προϊόντων καλύτερα θα καλυφθεί ε, μέσω των ε, συμφωνιών ε, αυτών. Και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο τελικά κατέληξε σε αυτή τη θέση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Πλέμπα. Η θέλεις να πεις δύο λόγια τελικά. Εγώ απλώς θέλω να επαναλάβω τις ευχαριστίες προς όλους και όλες τις ομάδες και ελπίζω ότι το Σεπτέμβριο θα ολοκληρώσουμε αυτή τη δουλειά. Ωραία. Ευχαριστώ Ιράτσε. Πάμε στο σημείο 15. Άλλο καλό νέο. Ο κανονισμός του Συμβουλίου για την ενιαία ενίσχυση προς στήριξη των αμπελοκαλλιοργητών. Και εδώ ο Ντόρφμαν είναι εισηγητή. 24 ε, Ιουλίου είχαμε τρίλογο στο Στρασβούργο και πήγε μια χαρά. Και καταλήξαμε σε μια συμφωνία σε όλες σχεδόν τις τροπολογίες της ε, Κόμαγκρη. Ο Χέρμπερτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, όντως έτσι είναι η κατάσταση. Αυτή η έκθεση είναι η πρώτη έκθεση του πακέτου της μεταρρύθμισης της γεωργίας που είναι μέρος των εθνικών φακέλων και καταρχήν σαν εισηγητής θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στη συζήτηση αυτή τις προηγούμενες εβδομάδες ε, όπως άλλωστε και τους συνεργάτες στη γραμματεία σε την ψηφοφορία που είχαμε στην Επιτροπή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροποποιήθηκε σε ορισμένα σημεία ε, και ε, αναρωτηθήκαμε αν τα εθνικά, η εθνική ε, φάκελη θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις άμεσες πληρωμές του πρώτου πληρώνω και θα αλλάξουν μετά από δύο χρόνια σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή ε, θα έπρεπε να αποφασίσουμε αμέσως για να έχουμε ένα ενδιάμεσο έτος ενώ ε, πρόκειται η τελική απόφαση να ληφθεί σε ένα χρόνο, δηλαδή το 2013. Πώς θα γινόταν δηλαδή μια καλύτερη προσαρμογή και ένας καλύτερος ο συντονισμό με τις υπόλοιπε πτυχές της μεταρρύθμισης αυτής ε, στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα την περασμένη Τετάρτη έγινε ένας τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου ουσιαστικά όλες οι τροπολογίες τις οποίες είχαμε υποβάλει στο Συμβούλιο υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ορισμένες γλωσσικές αλλαγές και βελτιώσεις ε, ε, ορισμένων ενιών, δηλαδή ε, συμπλήρωσαν αυτά που είχαμε αποφασίσει και εδώ στην Επιτροπή. Σχετικά με την τροπολογία της κυρίας Λούλινγκ, όπου ελέγεται ότι οι πόροι αυτοί από τους εθνικούς φακέλους δεν αποτελούν μέρος της συγκλήσεως μεταξύ των κρατών και δεν έπρεπε να αποτελούν μέρος της συγκλήσεως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο διότι η κατανομή των πόρων στα κράτη-μέλη θα επιτευχθεί πριν από τις αποφάσεις των μεμονωμένων χωρών σχετικά με το συγκεκριμένο κονδύλι του προϋπολογισμού. Δηλαδή θα προστεθεί στην ενιαία πληρωμή και γι' αυτό θα μπορέσει να γίνει μια ευρωπαϊκή κατανομή των πόρων ως εκ τούτου δεν μπορεί η σύγκληση να αποτελέσει μέρος των εθνικών φακέλων πληρωμής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, προσέθεσε μία παράγραφο που περιγράφει ακριβώς αυτή τη διαδικασία και όπιν αυτού περιτεύει αυτή η τροπολογία διότι τεχνικά δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει μέρος της συγκλήσεως αυτή η κατανομή. Ε, ελπίζω λοιπόν ότι το φθινόπωρο στην ψηφοφορία θα μπορέσουμε όντως τελικά σε πρώτη ανάγνωση και στο Συμβούλιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια να υιοθετήσουμε αυτή τη θέση και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Χέρμπερτ. Δύο σημαντικοί τρίλογοι που κατέληξαν ε, θετικά. Αν κανένας ε, δεν θέλει το λόγο και επειδή δεν έχουμε και εκπροσώπους της Κομισιόν, Ολοκληρώνουμε λοιπόν το 15. Και τώρα μισή ώρα διάλειμμα, 40 λεπτά καλύτερα, διότι στις 11 θα έρθει ο Σοφοκλής Αρετράρης, ο Κύπριος Υπουργός Γεωργίας, για να μας αναφέρει το πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας στις 11 παρα 5. Διάλειμμα. Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Αρχίζουμε. Αρχίζουμε καλωσορίζοντας θερμά τον νέο προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τον κύριο Σοφοκλή Αλετράρη, Υπουργό Γεωργίας που θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας σήμερα. Αγαπητέ Σοφοκλή, η Προεδρία σου είναι μία προεδρία που πέφτει σε μία σταυρική στιγμή της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Βρίσκεται στο μέσο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Σε μία φάση όπου η Επιτροπή μας επεξεργάζεται τις θέσεις της για διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Όπως γνωρίζεις, η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για τη μεταρρύθμιση είναι στις 13 Ιουλίου και έχουμε λάβει πάνω από 1.100 τροπολογίες. Ε, ελπίζω να συνεργαστούμε στενά για την ανταλλαγή πληροφόρησης και να κατανοήσουμε καλύτερα τις κοινέ θέσει του Συμβουλίου και της, Κομισ... της Επιτροπής μας για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Φυσικά όμως αγαπητέ Σοφοκλή υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα για τα οποία σίγουρα θα μας μιλήσεις και λέω επίσης ότι είχαμε μια πολύ καλή αρχή με την Κυπριακή Προεδρία διότι την προηγούμενη εβδομάδα το συζητήσαμε στις 4 Ιουλίου κιόλας ολοκληρώσαμε τον τρίλογο για το καθεστώς των άμεσων πληρωμών και το καθεστώς υποστήριξης των αμπελουργών. Σου δίνω το λόγο με ιδιαίτερη ικανοποίηση και σε καλωσορίζω θερμά και καλή επιτυχία για την Προεδρία σου. Σοφοκλή, έχεις το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι με μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση που σας παρουσιάζω σήμερα τις προτεραιότητες του Συμβουλίου στον τομέα της γεωργίας για τους επόμενους έξι μήνες. Η Κυπριακή Προεδρία προσβλέπει σε μια παραγωγική συνεργασία ανάμεσα στα δύο θεσμικά μας όργανα στο ίδιο θετικό πνεύμα που σημειώθηκε τους προηγούμενους έξι μήνες κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας. Κύριε Πρόεδρε, από τον Οκτώβρη του περασμένου χρόνου η συζήτηση των προτάσεων της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής του Επιτρόπου Σιόλου αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο συζήτησης τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο. Είμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση της αναδιαμόρφωσης της κοινή αγροτικής πολιτικής ώστε να απαντήσει στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων γεωργών, των πολιτών και των φορολογούμενων. Τα δύο θεσμικά μας όργανα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο καθορισμού των θέσεών τους όσον αφορά το πακέτο μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής. Στο Συμβούλιο έχουμε πετύχει ένα σημαντικό βήμα με την έκθεση προόδου που παρουσίασε η Δανική Προεδρία στα μέσα Ιουνίου. Στο Κοινοβούλιο έχετε επίσης προχωρήσει σημαντικά με την παρουσίαση των προσχεδίων εκθέσεων των αντίστοιχων εισηγητών σας, των αξιότιμων μελών του Κοινοβουλίου, Καπούλα Σάντος, Ταντάν και Λαβία θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόοδο της Επιτροπής σας και αναμένουμε να δούμε τις τελικές εκθέσεις αργότερα αυτό το χρόνο. Στο Συμβούλιο η Κυπριακή Προεδρία έχει ήδη ετοιμάσει ένα εντατικό χρονοδιάγραμμα συζητήσεων σε όλα τα επίπεδα. Στηριζόμενα στην έκθεση πρόοδου της Δανικής Προεδρίας θα προωθήσουμε την εργασία περαιτέρω ευελπιστώντας το ξεκαθάρισμα θέσεων του Συμβουλίου στα θέματα που εκκρεμούν. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί αρκετό έργο υψηλής ποιότητας, αλλά απομένουν ακόμα περισσότερα να γίνουν. Σε επίπεδο Υπουργών θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο μια πρώτη πολιτική συζήτηση για θέματα αγροτικής ανάπτυξης και κοινή οργάνωσης αγοράς. Επίσης έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω συζητήσεις για τις επόμενες συνόδους του Συμβουλίου. Στόχος μας είναι να πετύχουμε στο Συμβούλιο του Νοεμβρίου μια μερική γενική προσέγγιση η οποία θα αποτυπώνει για κάθε ένα από τα τέσσερα σχέδια κανονισμών το κέντρο βάρους στο Συμβούλιο. Αυτό θα διευκολύνει τις συζητήσεις στα θέματα της μεταρρύθμισης που είναι συνδεδεμένα με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θα συζητηθεί στο επίπεδο αρχικών κρατών. Ευελπιστούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνάντηση του Δεκέμβρη θα μπορέσει να κάνει αποφασιστική πρόοδο σε αυτά τα θέματα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συνεργασία μας με την Επιτροπή σας δεν μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για την στήριξη στους αμπελοκαλλιεργητές, καταφέραμε να φτάσουμε σε συμφωνία κατά τη διάρκεια του τριλόγου στο Στρασβούργο στις 4 Ιουλίου, την τέταρτη δηλαδή μέρα της Προεδρίας μας. Τώρα αναμένουμε την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση κατά τη σύνοδό της 10 με 13 Σεπτεμβρίου. Τώρα θέλω να αναφερθώ στη συμφωνία του μεταβατικού κανονισμού για τις άμεσες πληρωμές για τον οποίο η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση κατά τη Σύνοδο την περασμένη εβδομάδα. Λόγω της εξαίρετης μας συνεργασίας, οι δύο κανονισμοί, τόσο εκείνος για τη στήριξη στους αμπελοκαλλιεργητές, όσο και εκείνος της μεταβατικής περίοδου για τις άμεσες πληρωμές έχουν μεγάλες πιθανότητες να αρχίσει η εφαρμογή τους από την 1η Ιανουαρίου 2013 όπως έχει προγραμματιστεί. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μεμονωμένα. Ένας βιώσιμος, παραγωγικός και ανταγωνιστικός γεωργικός ευρωπαϊκός τομέας είναι σημαντικός για να ικανοποιήσει τις ανάγκες σε τρόφιμα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρειαζόμαστε όμως επίσης μια συλλογική και συνεχτική λύση στο πρόβλημα της επισητιστικής ανασφάλειας των τροφίμων διεθνώς. Με αυτή την έννοια τα πρότιμα τροφίμων COTEX Alimentarius είναι μεγάλη σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες καθότι έχουν ως στόχο να εγγυηθούν την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και τις ορθές πρακτικές στο εμπόριο τροφίμων. Τα, πρότιμα, τα πρότυπα τροφίμων του Κότεξ σχετίζονται άμεσα με το διεθνές εμπόριο τροφίμων και κατά συνέπεια έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το πρώτο εξάμεινο του 2012 η Δανική Προεδρία επιτέλεσε θαυμάσια εργασία με δραστηριότητες σχετικές με τα διεθνή πρότυπα και κατάφερε να αυξήσει στο μέγιστο βαθμό την επιρροή της στο φορέα αυτό. Λόγω των περιορισμένων πόρων, η Κύπρος ζήτησε υποστήριξη από τη Δανική Προεδρία, η οποία αποδέχτηκε να συνεχίσει το έργο αυτό και κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2012. Είμαι βέβαιος ότι η Δανική ομάδα θα συνεχίσει να υπερασπίσεται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίζει την διατήρηση των υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών στα τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχομαι τώρα σε ένα σημαντικό οριζόντιο θέμα που είναι η ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Με αυτό ενώ την επανεξέταση των προτάσεων της Επιτροπής για τη διαφοροποίηση ανάμεσα στη βασική πράξη της κατεξουσιοδότηση πράξης και τις εκτελεστικές πράξεις. Πρόσφατα, τα θεσμικά μας όργανα έχουν αρχίσει ανεπίσημους τριλόγους για διάφορα θέματα. Αυτά περιλαμβάνουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα μικρά νησιά του Αιγαίου και την βιολογική καλλιέργεια. Είμαι της άποψης ότι με την 20 εμπειρία τα θεσμικά μας όργανα έχουν σαφή αντίληψη αυτού του σημαντικού θεσμικού ζητήματος. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στη δημιουργία ομοιόμορφων συνθήκων εφαρμογής για όλες τις πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Όσον αφορά τώρα τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, πραγματοποιήθηκε τρίλογος κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας, κατά τον οποίον τόσο το Ευρωκοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο κατάφεραν να προσδιορίσουν καλύτερα τα, ζητήματα που διακυβεύονται. Ωστόσο, μετά από αυτόν τον τρίλογο δεν έγινε κατορθωτή οποιαδήποτε πρόοδος στο Συμβούλιο. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια σε αυτό το θέμα και να το ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, παράλληλα με τις συζητήσεις για το φάκελο για τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Για την βιολογική καλλιέργεια αναγνωρίζω τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε η Δανική Προεδρία στο θέμα αυτό. Η προκάτοχός μου διερεύνησε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω τρυπών, τριών άτυπων τριλόγων πιθανούς τρόπους για κοινό συμβιβασμό σε πρώτη ανάγνωση παρά το ότι σχεδόν όλα τα θέματα είχαν επιληθεί, παρατηρήθηκα μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων όσον αφορά τα δύο άρθρα. Ωστόσο, στο στάδιο αυτό, παρά το ότι η Δανική Προεδρία υπέβαλε συμβιβαστικές λύσεις, δεν στάθηκε δυστυχώς δυνατό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δεχθεί την προσφορά αυτή σε πρώτη ανάγνωση. Πέρασαν 18 μήνες από την υποβολή της σχετικής πρότασης από την Επιτροπή και πρέπει να αναζητήσουμε ειλικρινά και από κοινού ένα τρόπο να προχωρήσουμε. Σας διαβεβαιώ ότι η Κυπριακή Προεδρία είναι πλήρως δεσμευμένη στο να πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο σε όλους τους σχετικούς με την ευθυγράμμιση φακέλους σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε όλοι επιτυχή και εφαρμόσιμα αποτελέσματα στους φακέλους αυτούς. Όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας, όπως γνωρίζετε, η θέση μας είναι σαφής σε όλα σχεδόν τα σημεία, συμπεριλαμβανόμενης και της διαγραφής της πρότασης για γενικό κανόνα εμπορίου. Για τα δύο εναπομείναντα ανοιχτά ζητήματα, δηλαδή το πεδίο συγκεκριμένων κανόνων εμπορίας και την υποχρεωτική αναγραφή του τόπου γεωργικής παραγωγής, παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε την εργασία παράλληλα με το θέμα του ελέγχου των πολίσεων. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα εξετάσουμε τα θέματα αυτά στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η πρόθεση των γεωργικών προϊόντων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα και του τομέα επεξεργασίας τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την επιτυχία της μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής. Για τον λόγο αυτό, η Προεδρία υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία μεταρρύθμισης της πολιτικής πρόθεσης που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2011. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται ήδη στη δεύτερη της φάση μετά την έκδοση εκ μέρους της Επιτροπής στις 30 Μαρτίου 2012 της ανακοίνωσης με θέμα ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και πρόθεσή τους. Προσβλέπουμε στην έκφαση της συζήτησης που ξεκίνησε με την έκδοση της ανακοίνωσης και ιδίως στις νομοθετικές πράξεις που θα παρουσιάσει η Επιτροπή μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου. Όσον αφορά τον τομέα της υγείας των ζώων, της ζωικής παραγωγής και των τροφίμων ζωικής προέλευσης, αναμένουμε από την Επιτροπή να υποβάλει μια σειρά σημαντικών νομοθετικών πράξεων στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Η πρώτη από αυτές είναι η πρόταση για αναδιατύπωση της ζωοτεχνικής νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διατάξεις αυτές είναι για την ώρα διεσπαρμένες σε 11 πράξεις του Συμβουλίου, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους σε διάφορα ζητήματα λεπτομεριών. Η τελική προσπάθεια της Επιτροπής θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της συνοχής τους, την πλήρη εφαρμογή τους, την προσβασιμότητά τους και την νομική τους σαφήνεια. Σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισαβόνας, η νομοθετική πρόταση εμπίπτει στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, δηλαδή της συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η δεύτερη πρόταση αφορά τον τομέα της παραγωγής τροφίμων, δηλαδή τους κανόνες για υγιεινή παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών. Η νομοθεσία αυτή που υιοθετήθηκε το 2004 και είναι γνωστή ως δέσμη υγιεινής, αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της πολιτικής από το αγρόκτημα στο τραπέζι χάρη στην καινοτόμο φύση της προσέγγισης αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζήτησαν όπως η Επιτροπή υποβάλει σχετική έκθεση μόλις τρία χρόνια μετά την εφαρμογή της. Η έκθεση με τις εμπειρίες των πρώτων χρόνων εφαρμογής υποβλήθηκε το 2009 και εξετάστηκε τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει των σχολείων μας και πρόσθετων διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους παράγοντες αναμένεται σύντομα κατάθεση πρότασης αναθεώρησης. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε αναμένεται υποβολή της εντός του Οκτωβρίου και ελπίζουμε πως η νέα πρόταση θα είναι απλούστερη και με ξεκάθαρες πρόνοιες οι οποίες θα στοχεύουν αφενός στη μείωση του διοικητικού φόρτου και αφετέρου στη διατήρηση του ψηλού επίπεδου προστασίας του καταναλωτή. Η τρίτη πρόταση που αναμένουμε είναι εκείνη η πιο φιλόδοξη. Πρόκειται για το σχέδιο νέου και ολοκληρωμένου νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων αναμένεται να υποβληθεί ως μέρος μιας σειράς προτάσεων που θα περιλαμβάνουν επίσης φυτογιονομικά θέματα και σπόρους προσπορά. Με αυτή την νομοθεσία στοχεύεται μια πολύ απλή εφαρμογή του γενικού εμβλήματος της στρατηγικής για την υγεία των ζώων η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία παρά το ότι, όπως έχω πληροφορηθεί, ενδεχομένως να υπάρξει καθυστέρηση στην υποβολή του σημαντικού αυτού πακέτου νομοθετικών προτάσεων, ειλικρινά ευελπιστώ όπως αυτό παρουσιαστεί τελικά από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, προκειμένου τα δύο θεσμικά όργανα να αρχίσουν την επεξεργασία του κειμένου προς το συμφέρον των Ευρωπαίων Γεωργών και Χτινοτρόφων των λοιπόν φορέων που εμπλέκονται στην τροφική αλυσίδα και κατ' επέκταση των ιδίων των καταναλωτών. Όπως η Ιδανική Προεδρία με τις προτάσεις για την ηλεκτρονική σήμανση των βοηδών, την προαιρετική σήμανση του βόηου κρέατος και τη διακίνηση των κατοικίδιων ζώων, έτσι και η Προεδρία μας αναμένει ότι θα εργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα σε ένα θετικό και επικοδομητικό πνεύμα ώστε να οδηγήσει σε κοινέ αποφάσεις. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω διαβεβαιώνοντάς σας ότι η Κυπριακή Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί τους προσεχούς μήνες για να εξασφαλίσει τον ειλικρινή διάλογο ανάμεσα στα θεσμικά μας όργανα, ο οποίος θα αποτελεί ισχυρό θεμέλιο για τις φιλόδοξες και ισορροπημένες συμφωνίες το δεύτερο εξάμενο του 2012 και πέραν από αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρε, θα χαρώ να δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ αγαπητέ Σοφοκλή, είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που όπως είπαμε και πριν έχει ξεκινήσει ήδη με απτά αποτελέσματα. Χάρηκα που άκουσα για το πώς προσδίδει ιδιαίτερη σημασία η Κυπριακή Προεδρία στην προσαρμογή των ευρωπαϊκών ε, διατάξεων και νομοθεσίας στη συνθήκη της Λισαβόνας. Όπως γνωρίζεις, εμείς εργαστήκαμε σκληρά και στις τρεις προηγούμενες προεδρίες, Ουγγρική, Πολωνική και Δανική, δεν καταφέραμε να βρούμε συμφωνία. Ελπίζω να, να προχωρήσουμε η Κυπριακή Προεδρία. Είναι πολύ σημαντικά θέματα. Στο προηγούμενο Στρασβούργο είχαμε ψηφοφορία στην Ολομέλεια για, τους, ε, για τα πρώτα έξι κείμενα προσαρμογής στη Λισαβόνα και όπως ε, γνωρίζεις, ο συσχετισμός ε, στην Ολομέλεια ήταν πάνω από 95% υπέρ, δηλαδή τεράστια υποστήριξη στη δουλειά αυτής της Επιτροπής. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας είπες. Έχουν εγγραφεί διάφοροι συνάδελφοι, ο Άλμπερτ και μετά ο Λουίς Κάπουλα Σάντος. Ο Άλμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας και αν σήμερα δεν παρίστανται πολλοί συνάδελφοι κύριε Υπουργέ, αυτό δεν οφείλεται στο ότι αδιαφορούν, αλλά δυστυχώς αυτή την εβδομάδα τελειώνει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και βλέπετε ότι πολλοί συνάδελφοι ε, υπογράφουν ακόμη τις τροπολογίες Έχω και εγώ 57 τροπολογίες ε, τις οποίες υπέγραψα μόνο για το δεύτερο πυλώνα. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αντιμετωπίζονται ε, διάφορα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι χρέος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βελτιώσει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία ερώτηση κύριε Πρόεδρε από την ανακοίνωση τύπου της συνεδριάσεως του Συμβουλίου με ενόχλησε ότι η Κύπριος είναι η μόνη η οποία χαιρέτησε τις νομοθετικές προτάσεις όπως υπευλήθησαν ενώ όλες οι άλλες χώρες ε, κάτι κατέκριναν. Τι σας οδήγησε στο να ε, επικροτήσετε αυτές τις προτάσεις διότι εμείς έχουμε ορισμένες ε, ε, απόψεις οι οποίες θεωρούν ότι ε, δεν συνάδει να επικροτεί κανείς όλες αυτές τις αποφάσεις είναι πολύ σημαντικό το εξάμεινο της Προεδρίας σας για την γεωργική πολιτική μετά το 2014 είμαστε στο σημείο όπου θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις και για να μπορέσουμε εγκαίρως να εφαρμόσουμε όλο το πακέτο θα χρειαστεί και εδώ σας ε, ε, ζητώ συγγνώμη γιατί άργησα και δεν ξέρω αν θίξατε ήδη το θέμα ε, θα ήθελα να μου πείτε σχετικά με το πακέτο πώς αξιολογείται τι την ε, προώθηση της χρηματοδότησης για μετά το 2014 μέσα στην Προεδρία σας γιατί τώρα θα συζητήσουμε για τα νομοθετικές προτάσεις θα ψηφίσουμε αλλά μπορούμε να ψηφίσουμε τελεσίδικα κύριε Υπουργέ μόνο όταν θα ξέρουμε πώς ε, θα διεξαχθεί από το 2014 η χρηματοδότηση γιατί δεν είμαι από τους πολιτικούς που μπορούν να χαρίζουν έτσι υποσχέσεις αλλά επειδή είμαι βαβαρός γεωργός ένα έχω υποσχεθεί στους γεωργούς μου ότι η γεωργική πολιτική μετά το 2014 όπου θα υπάρχουν 20% λιγότερη χρηματοδότηση και 30% περισσότερη γραφειοκρατία είναι κάτι που δεν θα δεχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα μπορούμε να σας πούμε τι μπορεί να δεχθούν και να ανεχθούν οι γεωργοί μας και να είναι σαφές. Αυτό το οποίο πρότεινε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαίνει ότι για τους γεωργούς ε, θα μειωθούν σημαντικά οι πόροι διότι αυτά τα οποία θα γίνουν παραδείγματο χάρη η αφαίρεση 7% από τις εκτάσεις παραγωγής θα οδηγήσουν σε μία αύξηση του κόστους και αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε και να διατηρήσουμε την ε, ε, ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων γεωργών πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Οι γεωργοί κάνουν προσπάθειες αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνονται παράλογες προτάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν την παραγωγή στην Ευρώπη σε μία κατιούσα. Θα πρέπει να θρέψουμε τους Ευρωπαίους και η Ευρώπη έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει μία ποιοτική διατροφή και μπορώ να σας πω ότι θα συνεργαστούμε εν ονόματι της πολιτικής μας ομάδας πολύ καλά μαζί και έχουμε δίπλα σας ένα εκπρόσωπο της πολιτικής σας ομάδος ο οποίος θα σας στηρίξει και προσβλέπουμε σε μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ Άλμπερτ. Το λόγο έχει ο Λουίς Κάπολος Σάντος παρακαλώ. Λουίς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω βεβαίως ε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου στην Επιτροπή μας ε, και σας εύχομαι τα καλύτερα, τις ειλικρινέστερες ευχές μου για καλή επιτυχία στη διάρκεια του εξαμήνου σας. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ε, ότι εκτιμώ την επιθυμία σας, την βούληση τη δική σας αλλά και των πολιτικών και τεχνοκρατών συνεργατών σας σχετικά με τις γενικές κατευθύνσεις ε, που θα ακολουθήσετε. Έχουμε ήδη συναντηθεί και στα πλαίσια της Δανικής Προεδρίας και γνωρίζω ότι επιθυμείτε πραγματικά σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να εγκαταστήσετε έναν καλό διάλογο και μια συνεκτική πολιτική και επομένως χαίρομαι ιδιαίτερως για, την, ε, για τις διεργασίες σε αυτές και για την προσέγγιση σας που δείχνουν πολύ καλή θέληση. Όσον αφορά τώρα τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας, θα συμφωνήσω φυσικά η Κυπριακή Προεδρία επιθυμεί να εστιαστεί στους ε, κανονισμούς που δημιουργούν πρόβλημα τούτη τη στιγμή. Είναι σαφές ότι οι διαπραγματεύσεις ε, ε, δεν θα είναι εύκολες. Είναι φυσικό του λεχθέντος όμως. Εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Το θέμα δηλαδή της χρηματοδότησης της ΚΑΠ. Πιστεύω ότι με πολιτικούς όρους θα ήταν θετικό, θα ήταν καλό να βρεθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα πολιτική συμφωνία όσον αφορά αυτό το αμφιλεγόμενο πολιτικό ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα της ε, αναδιανομής. Αν μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο σημείο αυτό, θα ήταν πραγματικά εξαιρετικό πράγμα, γιατί διαφορετικά ε, οι διαπραγματεύσεις θα υποφέρουν, πιστεύω, από αυτό το πρόβλημα. Γνωρίζετε τη θέση μας βεβαίως πάνω σε αυτό το ευαίσθητο θέμα ε, και ε, θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν να προσθέσετε την προτεραιότητα αυτή στον κατάλογο των προτεραιοτήτων ε, που μας αναφέρατε. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε μαζί να προχωρήσουμε και στο τέλος της Προεδρίας θα είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι τώρα. Ευχαριστώ ο Μισελ Ντοντά και ο Τζοβάνι Λαβία. Μισελ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ και αναπτύξατε ένα πρόγραμμα ε, στο οποίο μπορούμε να διακρίνουμε την ε, ε, σαφή σας βούληση να προωθήσετε θέματα τα οποία μας είναι ιδιαίτερος προσφυλή. Ε, όσον αφορά την ΚΟΑ, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της ευθυγράμμισης. Εδώ και πολλούς μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθορίσει κάποιες γραμμές. Οι διαπραγματευτές μας έδειξαν μεγάλη αποφασιστικότητα. Όπως είπε και ο Πρόεδρος προλίγου, το Κοινοβούλιο ψήφισε σχεδόν ομόφωνα σε πρώτη ανάγκη την κατευθυντήρια γραμμή μας και επομένως βασιζόμαστε απάνω σας κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου έτσι ώστε να προωθήσετε τη σκέψη και των συναδέλφων σας στα πλαίσια της συνθήκης του, της Ελισαβόνας γιατί πλέον το Κοινοβούλιο είναι συν, ε, ε, ε, είναι συν είναι συν νομοθέτης και επομένως συμμετέχει στην ε, συναπόφαση ε, ε, πραγματικά και ουσιαστικά και όχι έτσι για τους τύπους μονάχα. Μετά την τελευταία μεταρρύθμιση της ΕΚΑΠ έχουν υπάρξει βαθιές αλλαγές στον κόσμο. Διαπιστώνει κανείς ότι η απλή διαχείριση των αγορών δεν είναι ικανή έτσι ώστε να διασφαλιστεί αφενός η ορατότητα και ταυτοχρόνως η ασφάλεια και η εγγύηση των παραγωγών μας πολλές μεγάλες χώρες επαναδιατυπώνουν την γεωργική τους πολιτική συμπεριλαμβανομένων και χωρών οι οποίες μέχρι χτες ε, θεωρούν το αναπτυσσόμενες χώρες και οι οποίες σήμερα είναι οι άμεση ανταγωνιστές μας σε πολλές αγορές. Βραζιλία ας πούμε για παράδειγμα. Η Βραζιλία πρόσφατα αποφάσισε μια πολύ σημαντική αύξηση ε, του ε, γεωργικού της προϋπολογισμού. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, όχι μονάχα τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία τα οποία μας γνωστοποιήθηκαν ε, ε, δίνουν πολύ αυξημένα ε, αριθμητικά στοιχεία, αλλά τα, οι Ηνωμένε Πολιτείε επαναδιατυπώνουν, τροποποιούν ε, ε, το σύστημα επιδοτήσεων υπέρ των γεωργών. Είναι παράδοξο λοιπόν που τούτη τη στιγμή ακριβώς η Ευρωπαϊκή, Επιτροπή, η, συγγνώμη, Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει να αφήσει στην τύχη της ε, την διαχείριση των αγορών που αφενός ήταν ε, θέμα προστασίας των γεωργών αλλά αφετέρου προεβλέπεται από τις συνθήκες ακριβώς με στόχο την προστασία των γεωργών. Είδαμε μεγάλη πτυτικότητα, μεγάλη ε, ε, τροποποίηση των ε, τιμών που δεν συνδέονται πλέον με το κόστος παραγωγής. Βλέπουμε ότι τελικά αυτοί οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν μικρότερη αγοραστική δύναμη είναι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν πρώτοι. Βλέπετε τι έγινε με την κρίση του γάλακτος που οφείλεται στην έκρηξη των τιμών σε μερικά μεταποιημένα προϊόντα, τα οποία, η οποία οδήγησε στου, τους ε, ε, καταναλωτές να αλλάξουν τον τρόπο των παραδοσιακών, με τον οποίο έκαναν τις αγορές τους, τον παραδοσιακό τρόπο κατανάλωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μεταφέρετε στο σύνολο των συναδέλφων σας στο, στο, στο Συμβούλιο ότι δεν μπορεί να είναι μοναχικός καβαλάρης ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν μπορούμε να μείνουμε στις αρχές του 20ου αιώνα. Είμαστε στον 21ο. Ευχαριστώ Μισελ. Ο Τζοβάνι Λαβία. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την ε, Προεδρία για τις ε, πληροφορίες που μας έδωσε σχετικά με το πρόγραμμα του εξαμήνου για το Συμβούλιο ε, Γεωργίας. Θέλω να σταθώ σε δύο-τρία σημεία που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη δουλειά μας σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Το πρώτο δεν είναι άμεση αρμοδιότητα του κυρίου Αλετράρη, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να ασκήσει την επιρροή του στο Συμβούλιο για να επιταχύνει την εξέταση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Εμείς είπαμε σε αυτήν την Επιτροπή ότι δεν θα έχουμε την τελική ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο αλλά δεν έχουμε μία απόφαση για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι φήμες που κυκλοφορούν από την ομάδα επαφής μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου δεν είναι και πολύ καλές φήμες. Διότι δεν ήταν ευτυχής η απόλυξη της ε, δανικής προεδρίας. Σίγουρα είχαμε συζήτηση και αντιπαράθεση, αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε ένα διαπραγματεύσει, μια βάση διαπραγμάτευσης για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε βάζοντας νούμερα και μεγέθη. Βλέπουμε επίσης ότι ε, στο Συμβούλιο οικονομικών υπάρχει δυσκολία να εξετάσουν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και όλα τα μέτρα που αφορά στη χρηματοδότηση της Ένωσης. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα θέματα, διότι υποσκάπτουν τις προθεσμίες για τις μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ. Χρειαζόμαστε μια τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουμε έγκαιρα να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεύτερο που θα ήθελα να θίξω είναι αυτό το οποίο εσείς λαμπρά αναφέρατε για την ευθυγράμμιση. Για να είμαστε όμως ειλικρινείς, η σχέση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για την συνθήκη της Λισαβόνας δεν λειτουργήσε με τον καλύτερο τρόπο. Πέρασαν 18 μήνες και δεν καταλήξαμε ακόμη σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Κατά την Πολωνική Προεδρία είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις για να καταλήξουμε σε, μια, σε ένα αποτέλεσμα για την ευθυγράμμιση των, με την πολιτική της Λισαβόνας, στην Δανέζικη Προεδρία για τα γεωργικά έχουμε σταματήσει και δεν καταφέραμε να βρούμε μια λύση. Αυτό θα έχει, φαντάζομαι, επιπτώσεις ε, στο χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, διότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τροπολογίες που θέτουν ε, που τίθενται από το Κοινοβούλιο αφορούν στην ευθυγράμμιση. Πέρα από τα ειδικά και τεχνικά θέματα που αφορούν στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, θα πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε και τα προβλήματα ευθυγράμμισης που θα μπορούσαμε κάλλιστα να τα είχαμε λύσει από πριν και να τα είχαμε ξεφορτωθεί. Όμως το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε δώσει μας εξαντλεί. Διότι τελικά οι τροπολογίες πέρα από τα τεχνικά ζητήματα αφορούν και στην Λισαβόνα. Για τον οριζόντιο κανονισμό τώρα. Το Κοινοβούλιο μέσω εμού, ως εισηγητή, άρχισε να εκφράζει ορισμένες θέσεις που απορρέουν από τις συζητήσεις μέσα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή μας. Εμείς ψηφίσαμε την έκθεση Λάιον και μετά στην έκθεση ΔΕΣ εκφράσαμε έντονα την ανάγκη απλούστευσης. Πολλές τροπολογίες λοιπόν αφορούν στην απλούστευση, στην δημιουργία επίσης ενός συστήματος σήμανσης συναγερμού που να μειώνει το ρίσκο της κύρωσης του Γιωργού από λάθη που είναι περισσότερο ατυχήματα και όχι εκ Και για το θέμα των κυρώσεων, και αυτό το εκφράζουμε έντονα εδώ στις συζητήσεις της Επιτροπής μας, ότι Δεν θα, πρέπει να, θα πρέπει να υπάρχει ένα έντονο ε, στοιχείο ε, επιβολής κυρώσεων ε, για τον Γεωργό πρέπει να υπάρχει μία διάκριση μεταξύ του ευκαιριακού λάφους της παράληψης έναντι του νόμου από ότι η εκπροθρέσεως απάτη πρέπει να υπάρχει διάκριση αυτό το τυχαίο λάθος πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Αυτά θέλω να υποβάλω στην προσοχή σας και θα ήθελα η Προεδρία να υποστηρίξει τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ Τζοβάνι. Τελειώσαμε με τους τρεις εισηγητές και τους δύο συντονιστές. Τώρα ο Αντιπρόεδρος, κύριος Παπαστάμκος. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τον Υπουργό, τον κύριο Λετράρη, για την εδώ παρουσία του. Προσυπογράφω πλήρως τα όσα είπε ο συντονιστής του ΕΛΚΟ, ο κύριος ε, Άλμπερτ Ντες, ότι θέλουμε μια ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική, λιγότερο γραφειοκρατική και με αφορμή αυτό το λιγότερο γραφειοκρατική κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να πάρετε μια πρωτοβουλία έστω σε πρώτο στάδιο, να θέσετε τις βάσεις, για να, ούτως ώστε να καταστεί στο εγγύς μέλλον η κοινή αγροτική πολιτική η πιο απλουστευμένη κατά την εφαρμογή της πολιτική. Συμφωνώ επίσης με όσα είπε ο κύριος Λαβία για την ευθυγράμμιση και με αφορμή της παρατηρήσεων για την ευθυγράμμιση ένα θέμα που είναι εδώ και 18 μήνες στο τραπέζι των διαθεσμικών συζητήσεων, ξέρετε πρέπει να γίνει σαφές ότι η ευθυγράμμιση δεν είναι θέμα διαθεσμικής κουλτούρας, διαθεσμικών προδιαθέσεων, αλλά είναι θέμα επιβαλόμενης διαθεσμικής συνεργασίας. Είναι θέμα διαθεσμικών διευθετήσεων που προνοούνται ήδη και πρέπει να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Ο κ. Νταντέν επίση έθιξε το θέμα των εξωτερικών πτυχών τη κοινή αγροτική πολιτική. Πάρα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα. Δεν θα επεκταθώ επί του παρόντο. Αλλά θέλω να σα πω κάτι το οποίο βίωσα χθε το βράδυ. Παρέθεσα δείπνο με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Παϊκού Κοινοβουλίου προ τον Πρόεδρο τη Βουλή τη Νέα Ζηλανδία και στην αντιπροσωπεία. Έχουμε πολύ φιλική προδιάθεση και έναντι τη Νέα Ζηλανδία και έναντι τη Αυστραλία διεπίστωσα και πρώτο, μάλλον πριν την διαπίστωσή μου, το πρώτο εξαγωγικό προϊόν που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κρασί και οι δύο χώρες ως γνωστόν. Διεπίστωσα ότι στη Νέα Ζηλανδία, λέω, πολύ φιλική φίλη χώρα, δεν θα βρεις ευρωπαϊκό κρασί να παραγγείλεις ε, σε κανένα εστιατόριο. Θα μου πείτε αυτό είναι καταναλωτικός εθνοκεντρισμός δεν θέλω να το σχολιάσει περαιτέρω. Έχω τα καλύτερα αισθήματα απέναντι σε αυτέ τι δύο χώρε. Ε, Βεβαίω και κλείνω για τι εξωτερικέ πτυχέ. Θα πρέπει και αναδυόμενε οικονομίε θα πρέπει να λάβουν τι ευθύνε στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη που πρέπει να πληρώνει με συνεχείς παραχωρήσει στο γεωργικό τομέα. Κύριε Πρόεδρε, σα θυμάται το γεγονός ότι ήσταν εδώ παρόν τις εργασίες της Επιτροπής Γεωργίας πολύ πριν αναλάβει η Κυπριακή Προεδρία τη σκητάλη για το, επόμενο, για το τρέχον εξάμεινο. Σας θυμά το γεγονός ότι τονίσατε τη συνέχεια. Δανική Προεδρία, συνεχίζει η Κυπριακή Προεδρία και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, τρέχουσα μια αποτελεσματική πολιτική διαχείριση, την οποία έχετε ήδη να επιδείξετε όπως πολύ σωστά είπατε, ε, δείγματα γραφής. Και πιστεύω απόλυτα, και αυτό το διαπιστώνετε και σήμερα, ότι είστε Προεδρία της διαβούλευσης, του διαλόγου και μιας βαθιάς δημοκρατικής αντίληψης. Δεν τα λέω αυτά με όρους συναισθηματικής φόρτισης. Το πιστεύω βαθύτητα. Αλλά ο σεβασμός αυτόν το οποίο επιδεικνύεται απέναντι στον συνομοθέτη, που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει να είναι όπλο σας επιχείρημα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Ότι, α, στο τάδε θέμα η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι σύμμαχος επιτυχίας της Προεδρίας και όχι το, και όχι το ανάστροφο. Δηλαδή να έρχεστε εδώ και να λέτε «Α, το Συμβούλιο δεν το δέχεται αυτό». Και πιστεύω, διερμηνεύοντας και τη στάση όλων των μελών της Επιτροπής Γεωργίας, ότι ναι, κατά τη διάρκεια αυτής της εξάμηνης Προεδρίας θα είμαστε σύστοιχοι, αλληλέγγυοι για μια ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική η οποία ε, εξυπηρετεί ε, δημόσια αγαθά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλή επιτυχία, γόνιμη και δημιουργικό εξάμενο. Γόνιμη και δημιουργική προεδρία. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο κύριε, τον κύριο Παπαστάνκο, η Μάριον Μαγκίνες και μετά ο Αγνιού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου που ήρθε σήμερα εδώ πολλά υπόθηκαν σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Γι' αυτό εγώ θα πω πολύ λίγα ε, όσον αφορά το θέμα αυτό, γιατί υποστηρίζω αυτά που υπόθηκαν από τους προελέσαντες συναδέλφους. Όσον αφορά το προπολογισμό όμως, ε, η ε, γεωργή μας ήταν πάρα πολύ υπομονετική μαζί μας αλλά Τώρα με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, του ζητάμε ακόμα περισσότερα μέσω του πρασινίσματος. Ε, του ζητάμε περισσότερα λοιπόν, αλλά τους δίνουμε λιγότερα αυτή τη στιγμή τα αναλώσιμα προϊόντα διαρκώς ε, γίνονται πιο ακριβά ε, και ε, προβλήματα, κρίση οικονομική πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που έχετε στο Συμβούλιο έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα του σωστού προϋπολογισμού. Και θα έρθω σε αυτό που είπε και ο συνάδελφος Μισελ Νταντάν σχετικά με τον ρόλο, με τον, τρόπο συγγνώμη, με τον οποίο βλέπουν άλλοι παγκόσμιοι ε, τη ε, της ε, γεωργίας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. βεβαίω θα είμαστε στη διάθεσή σα να συνεργαστούμε για τι λεπτομέρειε τη μεταρρύθμισης. Ε, τώρα κάτι άλλο. Καλωσορίζω τα όσα είπατε για την ε, ευζοία των ζώων. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό η υγεία των ζώων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει άμεσο αντίκτυπο και στην υγεία ε, της ε, εκμετάλλευσης. Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σας. Επίσης ε, το ζήτημα της αυτάρκειας των, της, τροφής, της ζωικής τροφής έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα μεταλλαγμένα και θα έχουμε ακόμα περισσότερο μεγάλο πρόβλημα τη στιγμή που η Γεωργία και άλλοι μεγάλοι παίκτες ε, της παγκόσμιας σκηνής έχουν την διάθεση να αγοράζουν ε, τρόφιμα τα οποία δεν είναι ελεγμένα. Δεν είναι ελεγμένα όσον αφορά τις πρωτεΐνες, όσον αφορά την πρόληψη της σόγιας ε, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο φάκελο του Επιτρόπου κυρίου Ντάλη. Ε, επίσης ε, το θέμα των ηλεκτρονικών ενωτίων των προβάτων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις φάρμες, για τις αγρικίες, για τους κτηνοτρόφους μας. Χρειάζεται κάποια παρέμβαση και από εσά ναι, και ο ρόλο σα είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίω, όπω είπαν και οι άλλοι μου συνάδελφοι, πραγματικά θα συνεργαστείτε μαζί σα και θα συνεργαστούμε και εμεί μαζί σα και ελπίζω ότι αυτό το δεύτερο εξάμεινο αυτή τη Προεδρία θα είναι ε, ισχυρό εξάμεινο, έστω και αν ξεκινάμε έτσι μέσα στις καλοκαιρινές ε, διακοπές. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσετε, θα πρέπει να προχωρήσουν και οι μεταρρυθμίσεις του επόμενου έξι μήνε γιατί διαφορετικά δεν πιστεύω ότι το 14 την 1η Ιανουαρίου θα έχουμε πραγματικά τη μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μάριον. Άγνιου και μετά σε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά την εκλογή μου το 2009 μου είπαν ότι τα πράγματα τώρα κύριε Άγνιου είναι διαφορετικά. Ε, υπάρχει συν απόφαση και το Κοινοβούλιο είναι σημαντικός παίχτης. Και όμως καθόμαστε σήμερα εδώ, πρώτη συνάντηση με τη Νέα Κυπριακή Προεδρία και βλέπω 8 βουλευτές. Ενώ βλέπετε πόσο πολυπληθής είναι η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου, της Κομισιόν, Μα εκπλήσωμαι. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα σήμερα με τις τροπολογίες, αλλά θα μπορούσαν οι συνάδελφοι να σταματήσουν για λίγο ε, τη δουλειά για τις τροπολογίες και να έρθουν εδώ. Μα ακόμα και οι πράσινοι απουσιάζουν, αν είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, μην πάρετε προσωπικά το επόμενο σχόλιο μου, κυρία Ελεκτράρη. Ξέρετε ότι έχω σημαντικές επιφυλάξεις όσον αφορά μια μικρή χώρα που βρίσκεται στην άκρη, άκρη, άκρη της Μεσογείου και η οποία καλείται αυτή τη στιγμή να ε, προχωρήσει στην μεταρρύθμιση, να διαχειριστεί τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτιέμαι πόσο μπορούν να στηρίξουν οι ώμοι της Κύπρου. Αλλά βεβαίως είσαστε εδώ έτσι ώστε να μου αποδείξετε ότι λανθάνω, ότι κάνω λάθος και ότι εσείς μπορείτε να κάνετε πολλά τους επόμενους έξι μήνες. Ε, κοιτάξτε, όσον αφορά τις ε, ε, προεδρίες, ξέρουμε ότι είναι έξι μήνες για το πρώτο εξάμεινο, αλλά η δεύτερη προεδρία δεν είναι και κανονικό εξάμενο. Επομένως, εσείς θα πρέπει να βάλετε πολύ ψηλή ταχύτητα, έτσι ώστε το λίγο χρονικό διάστημα που έχετε μπροστά σας να καταφέρετε αυτά που πρέπει να καταφέρετε. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την πρόταση για το πρασίνισμα. Υπάρχουν τρία σκέλη ε, τα οποία αφορούν ε, τρία διαφορετικά πράγματα. Ε, βλέπω όμως ότι ο Επίτροπος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα αυτά, τον είδα σε ένα βίντεο, δεν απήντησε πολύ καθαρά και ε, κατάλαβα ότι είπε ότι τα περιβαλλοντικά προγράμματα θα πρέπει να αφορούν μονάχα τις επικεντρωμένες περιβαλλοντικές περιοχές. Ε, και είπε ναι, ναι, έτσι είναι, αλλά δεν το έχουμε δει γραπτά. Θα πρέπει να το δούμε και γραπτά. Ε, όσον αφορά τώρα τα EFA η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δηλαδή, η πραγματικότητα είναι ότι τα αναλώσιμα ακριβένουν μέρα με τη μέρα. Και φαίνεται ότι η απάντηση σε αυτό είναι εντάξει ας αφαιρέσουμε καλλιεργητική γη από την παραγωγή. Μα αυτό είναι τρελό, είναι παράλογο. Ο κύριος Καπουλασάντος ε, έφτασε σε κάποιο είδος ε, συμβιβασμού. Γιατί καμιά φορά το μη είναι βέλτιστον. Τι να κάνουμε. Είπε λοιπόν ε, είπε λοιπόν, γιατί οι ε, πρωτεϊνικές ας πούμε καλλιέργειες ε, να μην ε, μπουν σε περισσότερες ε, καλλιεργήσιμες περιοχές. Ναι, θα μπορούσε να είναι αυτό. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα και ο Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου γιατί ξέρετε δεν, δεν θα ε, λαδώσουμε εντό εισαγωγικών τους γεωργούς ε, με αυτές τις πρωτεϊνικές καλλιέργειες και εγώ γεωργός είμαι και εγώ ίδιος ε, αλλά ούτε την άλλη μεριά θα πρέπει να τους απειλούμε και να τους εκβιάζουμε. Όσον αφορά το τρίτο σημείο του πρασινίσματος, δηλαδή την διαφοροποίηση των συγκομιδών και αυτό των σοδιών και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εάν έχεις πάνω από 8 εκτάρια θα πρέπει να έχεις τρεις διαφορετικές οδιές. Αυτό είναι αυτό είναι παράλογο. Ε, καταλαβαίνετε ότι ε, όταν έχει κανείς μία μικρή εκμετάλλευση ε, θέλει ας πούμε ενδεχομένως τη μία χρονιά να βάλει μόνο κρυθάρι, την άλλη χρονιά να βάλει μόνο σίκαλι ε, και βεβαίως και είναι πιο αποτελεσματικός τρόπος παραγωγής και κερδίζεις χρόνο κτλ. Όσον αφορά τώρα τα λιβάδια ναι, εντάξει, μας λένε θέλουμε μια ευελιξία, άλλοι λένε όχι να έχουμε και λιβάδια. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ελπίζω ότι πραγματικά θα δείτε από πολύ κοντά αυτά τα τρία ζητήματα ε, τα οποία αναφέρω και να συμφωνήσω βέβαια και με την ε, Μαρία Μαγκίνες ε, η οποία είναι από την Ιρλανδία όσον αφορά τα ενότια των προβάτων, τη σήμαση των προβάτων είναι κάτι που μας χτυπάει και μας, μας πλήττει και μας πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συναδελφάγνιου. Πέρα από το πρόβλημα των τροπολογιών έχουμε και μία διαδήλωση σοφοκλή γαλακτοπαραγωγών και διάφοροι βουλευτές μας πήγαν να διαδηλώσουν, λυπούμε. Ο αντιπρόεδρος η και μετά ο Άλμπρεστ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύσκολη εποχή, πολύ δύσκολη, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό επιτρέπει, κύριε Πρόεδρε, να παρακολουθήσουμε από κοντά τις ε, ενέργειές σας και τις ε, δράσεις σας. Εγώ έτσι ακούγοντάς σας ε, λέω ότι θα, το προχώρημα της μεταρρύθμισης θα είναι ένα κανονικό, ένα νορμάλ προχώρημα και πρέπει να εξυπηρετήσει τους γεωργούς. Εγώ θα, εξηγήσω, θα ξεκινήσω με το θέμα του προϋπολογισμού. Δεν έχουμε τα παλιά επίπεδα προϋπολογισμού, λένε. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Απλώς οι γεωργοί των παλαιών χωρών θα λάβουν μικρότερες ενισχύσεις για τις περισσότερες που θα πρέπει να λάβουν οι γεωργοί που, γίναν, που μπήκαν στην Ένωση το 2004. Τώρα οι γεωργοί της παλιάς Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε δεν διατηρείται ο προπολογισμό στα επίπεδα και τους μπαίνει και η ιδέα ότι ορίστε βγάζουμε από τους μεν για να δώσουμε στους δε. δεν θα ήταν δύσκολο να καθησυχάσουμε τα πνεύματα γιατί θα πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα και να τα διευκρινίσουμε καλά. Υπάρχουν ένα σωρό συμβιβασμοί και υποχρεώσεις ε, πέφτουν ε, στην καμπούρα των γεωργών και η κλιματική αλλαγή αλλάζει πολλά πράγματα στη γεωργία. Και τελικά πολλές φορές εμείς εδώ ξεψυρίζουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά. Και ξεχνάμε το κλίμα, ξεχνάμε το θέμα της παραγωγής τροφίμων που είναι ο βασικός ρόλος των γεωργών. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε και μια ιδιαίτερη σημασία στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος πληρώνει όλες αυτές τις εξωτερικές σχέσεις. Σε ποιανού την καμπούρα πέφτει. Στους γιοργούς πέφτει. Πολλά προβλήματα λοιπόν. Το θέμα της διαχείρισης και των όρων, των συνθήκων των γιοργών. Θα ήθελα οι γιοργοί να έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Θα ήθελα να αναζωογονήσουμε την Ήπεθρο. Και εμείς βλέπουμε να ενισχύονται περιοχές εκείνες οι οποίες έχουν και το μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό και την περισσότερη απασχόληση. Αλλά γιατί έχουν την απασχόληση, γιατί έχουν πληθυσμό. Γιατί υπάρχει κόσμος που κατοικεί σε αυτές τις περιοχές. Τώρα, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν καλό είναι να έχουμε καλές σχέσεις εργασίας αν θέλουμε να καταλήξουμε κάπου. Οι Πολωνοί, οι Γεωργοί ενδιαφέρονται για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου λένε ότι θα πρέπει να αφιερώσετε εξίσου χρόνο για τους Γιοργούς όσο αφιερώνετε και για την ευημερία των ζώων. Αυτό μου λένε οι Πολωνοί Γιωργοί. Ευχαριστώ πολύ ο συνάδελφος Άλμπρεχτ και μετά απάντηση του Προέδρου. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον ε, κύριο Υπουργό, καθώς επίσης και την Κυπριακή Προεδρία. Ε, δείχνεται μεγάλη αποφασιστικότητα και αυτό μας ικανοποιεί. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές στα πλαίσια της ΚΑΠ. Αυτές οι περιοχές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να υπογραμμίσω λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, ο αντίκτυπος των, ε, ε, ε, των συμφωνιών με την, για, την, για τις μπανάνες με τις χώρες της Νότιας Αμερικής ήταν ένα σημαντικό ζήτημα στον τριμερή διάλογο. Πρέπει να ζητήσουμε οπωσδήποτε και αποζημίωση με κάποιο τρόπο για τους παραγωγούς μπανάνας. Επίσης θα πρέπει το πρόγραμμα να είναι πιο ε, αντιδραστικό εντός εισαγωγικών ε, ε, και εξηγούμε. Θα πρέπει κάθε φορά που γίνονται τροποποιήσεις των εμπορικών συμφωνιών ή κάποια τροποποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής θα πρέπει να γίνεται ανάλυση αντικτύπου. Αυτή η ανάλυση αντικτύπου και επιπτώσεων είναι απαραίτητη εάν θέλουμε τελικά τα προγράμματα να δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα αποφασιστικό, ε, αποφασιστική και σοβαρή σημασία, κυρίω για αυτέ τι ιδιαίτερα απομακρυσμένε περιοχέ. Επίση, να πω το εξή. Η Κυπριακή Προεδρία οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει μια έτσι ευαίσθητη κατάσταση. Το ανέφερε άλλωστε και ο πρόεδρο τη Επιτροπή μα όσον αφορά τον γαλακτοκομικό τομέα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί επανειλημμένα παρακολουθήσατε ε, την εξέλιξη της παραγωγής, παρακολουθήσατε τον φάκελο του γάλακτος. Το κόστος της παραγωγής είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ψηλό, ενώ οι τιμές πώληση είναι εξαιρετικά χαμηλές ε, και επομένως ε, αυτό εξηγεί βεβαίως την απόγνωση των παραγωγών που δεν θα μπορέσουν άλλωστε να κρατήσουν και πάρα πολύ, να επιβιώσουν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, πολλό δε μάλλον που διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν ανισορροπίες όσον αφορά τη γαλακτοκομική αλυσίδα. Και επομένως έχουμε πρόβλημα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ανισορροπίας, μεγάλο πρόβλημα ε, οικονομικό, πρόβλημα εισοδήματος κτλ. Επιμένω λοιπόν στο σημείο αυτό, αλλά βεβαίως σας εύχομαι καλή τύχη και καλή επιτυχία. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους και θα δώσω για μία ακόμα φορά στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τον Υπουργό κ. Σοφοκλή Αλετράρη, έτσι ώστε να απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων και να κάνει και τα τελευταία του ε, σχόλια. Καλή επιτυχία λοιπόν για μία ακόμα φορά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε, εμείς κυρίες και κύριοι, ως Κύπρος, χαιρετήσαμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαν μια καλή βάση για τις συζητήσεις που λογικά θα πρέπει να ακολουθήσουν και για το γεγονός ότι εμπεριέχουν μια καλή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Η, η Κυπριακή Προεδρία θα συνεργαστεί στενά με όλους τους φορείς ώστε οι τελικές αποφάσεις να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής των Ευρωπαίων πολιτών. Ειδικότερα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω τη σημασία που δίδομαι στην απλοποίηση και στη μείωση του διοικητικού κόστους, κάτι για το οποίο επιμένουμε πάρα πολύ. Γιατί ελέγχθηκε πολύ σωστά ότι ζητούμε περισσότερα από τους γεωργούς αλλά τους υποβάλλουμε σε περισσότερη γραφειοκρατία. Το θέμα τώρα του προϋπολογισμού, ναι, πιστεύουμε ότι ο ισορροπημένος προϋπολογισμός που θα επιτύχει μια ε, δίκαιη και ισότιμη κατανομή των πόρων τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και εντός του κάθε κράτους αποτελεί ύψης της σημασίας στόχο για μας. Πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, σκοπεύουμε να εξετάσουμε όλες τις πιθανές επιλογές. Ωστόσο, πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας ότι η κατανομή του προπολογισμού αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και οποιασδήποτε εισηγήσεις για την κατανομή των κοντιλιών θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις αυτές, συμβάλλοντας ακόμα και στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσής τους. Τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, που είναι υπεύθυνα για την Γεωργία, δεν συζήτησαν ακόμα το θέμα της κατανομής των πόρων και αναμένουν την απόφαση από το, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ μετά το 2014. Είναι σε γνώση του Συμβουλίου οι προτάσεις του εισηγητή του κυρίου Καπουλασάντος και ανυπομονούμε πραγματικά να συνεργαστούμε μαζί του αλλά και με την Επιτροπή σας κύριε Πρόεδρε στο πλαίσιο αυτού του θέματος σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Τώρα είναι αλήθεια και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας από τους μεγαλύτερους παίχτες στο διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται σημαντικά από τις εξελίξεις. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ θα πρέπει όλοι μας κύριε Πρόεδρε να συνεργαστούμε για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για σταθεροποίηση των αγορών και για αντιμετώπιση τυχών κρίσεων. Στις διεθνείς μας σχέσεις πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί αλλά και επιθετικοί όπου χρειάζεται για προάσπιση των συμφερόντων της Ένωσης. Σίγουρα δεν πρέπει να υποκύπτουμε στον πειρασμό του προστατευτισμού αλλά όντας ρεαλιστές και ταυτόχρονα καινοτόμοι θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τα ποιοτικά και άλλα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών παραγωγών. Ελέγχθηκε κύριε Πρόεδρε, σχολιάστηκε μάλλον το Νικό Box. αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, επηρεάζουν σημαντικά τις εξελίξεις σε όσον αφορά τη συζήτηση και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και η προϋπόθεσή μας είναι να εγκαθιδρύσουμε μια στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή σας παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις ώστε το μέτρο του δυνατού να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα. Είναι πράγματι γεγονός κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ότι στο λεγόμενο negotiating box για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει συμπεριληφθεί και ορισμένα επιμέρους θέματα γεωργικής πολιτικής τα οποία θεωρήθηκε ότι συνδέονται στενά με τα κύρια θέματα του προϋπολογισμού. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω ότι η Κυπριακή Προεδρία θα σεβαστεί πλήρως τα καθιερωμένα θεσμικά πλαίσια για τη συζήτηση των θεμάτων αυτών και για τη λήψη των τελικών αποφάσεων. Όσον αφορά τα θέματα του οριζόντιου κανονισμού, είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της Ιδανικής Προεδρίας το Συμβούλιο προχώρησε σε μια εντατική τεχνική εξέταση της πρότασης αυτής. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σε κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις αποτελεί μεταξύ άλλων ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της εργασίας. Σε αυτή τη βάση η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει να εργάζεται τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο και στοχεύει να πετύχει μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο μέχρι τον Νιόβρη ή τον Δεκέμβρη της φετινής χρονιάς. Να φέρθηκε από αρκετούς κύριε Πρόεδρε ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου με την συνθήκη της Λισαβόνας. Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούμε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ότι ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου είναι διακοσμητικός. Έχει ένα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την όλη φιλοσοφία της συναπόφασης και γιατί αναβαθμίζεται ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να νιώθουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται και λαμβάνουν υπόψη αυτούς που άμεσα τους εκπροσωπούν, δηλαδή τους Ευρωβουλευτές. Και εμείς το σεβόμαστε πλήρως κύριε Πρόεδρε Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα καθορίσει το συνολικό προϋπολογισμό της ΚΑΠ και την κατανομή στους δύο πυλώνες της μέχρι να ληφθούν ε, αποφάσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος στον τομέα της γεωργίας και η Κυπριακή Προεδρία έχει αναπροσαρμόσει τους συναφείς στόχους και το πρόγραμμά της. Σε καμιά περίπτωση η Κυπριακή Προεδρία δεν ευνοεί επιπλέον μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταλήξει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα προγραμματική περίοδο 14-20 θα πρέπει να μειωθούν ουσιαστικά, η Κυπριακή Προεδρία θα ζητήσει, όπως η ήδη αποφασιστήσα μείωση του προπολογισμού της ΚΑΠ, συναξιολογηθεί μαζί με άλλους ουσιώδεις παράγοντες. Τώρα για το πρασίνισμα της ΚΑΠ θέλω να αναφέρω ότι η Ιδανική Προεδρία έχει αφιερώσει σημαντικό χρόνο για τη συζήτηση του πρασινίσματος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποβάλει κάποιες προκαταρκτικές προτάσεις. Ως Κυπριακή Προεδρία αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη σημασία του θέματος και το γεγονός ότι ενδεχομένως να συνδέεται και με θέματα προπολογισμού. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοούμε με αυτό. Πρόθεσή μας είναι να στο κατάλληλο στάδιο να επανέλθουμε στο θέμα και δεν θα διστάσουμε να υποβάλουμε νέες ιδέες και προτάσεις λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τις θέσεις τις οποίες θα διαμορφώσει στο μεταξύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις νέες εισηγήσει που υπέβαλε τον περασμένο Μάιο έχει δείξει ένα πνεύμα συνδιαλλαγής και συναντήληψης. Δεν έχω καμιά αμφιβολία κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ότι με τη, με τη στενή συνεργασία όλων μας θα εξευρεθεί χρυσή τομή στο θέμα αυτό. αναφέρθηκε το θέμα των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το θέμα αυτό ως Προεδρία και σας διαβεβαιώνομαι ότι αναγνωρίζεται η σημαντικότητα των συγκεκριμένων μέτρων για την Γεωργία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που προκαλούνται από τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι απόμακρες περιοχές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και το πρόβλημα των Πανανών, στο οποίο αναφερθήκατε. Γνωρίζουμε ότι οι συζητήσεις επί της οριζόντιας συμφωνίας εναρμόνισης έχουν επιβραδυνθεί. Θα προσπαθήσουμε να επιφέρουμε σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό, στοχεύοντας σε μια προκαταρκτική συμφωνία μέχρι το τέλος του χρόνου. Για τον λόγο αυτό, προσβλέπουμε σε περαιτέρω συζήτηση των τροποποιήσεων της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου, την Επιτροπή σας δηλαδή. Παράλληλα, θα συναντηθούμε με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, έτσι ώστε οι λύσεις που θα προκύψουν να είναι αποδοτικές και εφαρμόσιμες. Αναφερθήκατε εσείς, κύριε Πρόεδρε, για την κρίση στο γάλα και για το ότι γίνεται κάποια διαμαρτυρία έξω από το κτίριο μας σήμερα. Θα πρέπει να αναφέρω ότι το Συμβούλιο παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση στην αγορά του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Να πω ότι το θέμα αυτό βρισκόταν στην ατσέντα στο τελευταίο Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο και ο Επίτροπος Σιόλος ανέλαβε να ενημερώσει τους υπουργούς την ερχόμενη Δευτέρα που θα έχουμε κύριε Πρόεδρε το Συμβούλιο Υπουργών για την όλη κατάσταση και τα μέτρα τα οποία προτίθεται να πάρει η Επιτροπή για να αντιμετώπιση το πρόβλημα εάν πράγματι επιβάλλεται. Πιστεύουμε εμείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση να αντιδρά έγκαιρα και έχει σημασία κύριε Πρόεδρε του έγκαιρα, έχοντας στη διάθεσή της ε, όλα τα αναγκαία εργαλεία για να αντιμετωπίζει παρόμοιες καταστάσεις, ειδικότερα όταν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό και ευρύτερο τομέα όπως ο βιομηχανικός. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπίζονται τα έκτακτα προβλήματα και διαταραχές στην αγορά, είτε αυτές οφείλονται σε απότομες αλλαγές στις τιμές, είτε πρόκειται για απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά που ανάφερα πριν λίγο κύριε Πρόεδρε θα συζητηθούν την ερχόμενη Δευτέρα κατά την πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου υπό την Προεδρία μου. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω ότι η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί το θέμα σαν προτεραιότητα και ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την σταθεροποίηση της αγοράς και την αντιμετώπιση των κρίσεων και θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν προς την κατεύθυνση αυτή. Κύριε Άκνιους, αυτή η απάντηση έρχεται σε σας. Πράγματι, η Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό κράτος με περιορισμένους πόρους και έχει μια μεγάλη ευθύνη. Αλλά πιστεύουμε, κύριε Άκνιος, ότι με τη σοβαρότητά μας, την υπευθυνότητά μας και την αποφασιστικότητά μας και τη σκληρή μας δουλειά θα αντεπεξέλθουμε της πρόκλησης. Μίστερ Κύριε Άγνιος, ε, είμαι σίγουρος ότι θα βγείτε λάθος τελικά. Ότι θα αποδειχθεί ότι έχετε λάθος στην εκτίμησή σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ αγαπητέ Σοφοκλή, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους. Ολοκληρώθηκε η πρωινή μας συνεδρίαση λοιπόν. 3 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στις 3 ακριβώς θα ξανασυναντηθούμε. Καλό, καλές διακοπές ε, και βεβαίως και καλή δουλειά όσον αφορά τις τροπολογίες σας. Μην το παρακάνετε όμως. Ευχαριστώ.